Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Και αν έχετε πηγαδάκια, παρακαλώ να τα ε, συνεχίσετε εκτός εθούσης. Έχουμε καθυστερήσει λίγο. Περίμενα τον εισηγητή για τον προπολογισμό. Δεν μπορεί να είναι εδώ όμω. Υπάρχει κάποιο εκπρόσωπο του ΕΛΚ για να ε, σχολιάσει εκ μέρου του. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 9 και 10 για τον προπολογισμό στην ημερήσια διάταξη. Και τα δύο θέματα είναι για τον προπολογισμό. Πριν όμως ψηφίσουμε για τις ε, τροπολογίες ε, για τον ε, προπολογισμό για το 2015, μπορούμε να συζητήσουμε τις γενικές κατευθύνσεις, προτεραιότητες και προκλήσεις και να δούμε κατά πόσον θα θέλαμε να τις συμπεριλάβουμε όλες αυτές στην γνωμοδότησή μας προς το ε, για τον προπολογισμό. Αυτό είναι μη νομοθετικό κείμενο που υποβάλλεται στην Επιτροπή Προπολογισμών για ε, προσανατολισμού πολιτική. Θα ετοιμάσουμε λοιπόν μια γνωμοδότηση την οποία θα αποστείλουμε στην Επιτροπή Προπολογισμών και το κείμενο το οποίο έχετε ενώπιον σα από πλευρά του κ. Ρούμπιχ είναι ένα σχέδιο γνωμοδότηση με τι προτάσει του το οποίο και θα συζητήσουμε και φυσικά η Επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει την πρόταση του κυρίου Ρούμπιχ. Θα γίνει λοιπόν η συζήτηση και από εκεί και πέρα θα σας πω την προθεσμία για τις ε, τροπολογίες για την ε, ε, γνωμοδότηση. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Στέρ, ο οποίος αντικαθιστά τον κύριο Ρούμπιχ που δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων εκτός Βρυξελών, ο συντάκτης της γνωμοδότησης, ο κύριος Ρούμπιχ, δυστυχώς δεν μπορεί να παραστεί στη σημερινή συνεδρίαση, αλλά μου ζήτησε να σας εξηγήσω κάποια από τα επιχειρήματα ε, τα οποία διέπουν τη γνωμοδότησή του και φυσικά να σας πει και σε γενικές ε, γραμμές ε, τι προτείνει για τον προϋπολογισμό του 2015. Όπως ήδη συζητήθηκε στην συνεδρίαση των συντονιστών της Επιτροπής Ανάπτυξης τον Ιούλιο, το επίπεδο των πληρωμών σε επίπεδο των δεσμεύσεων είναι πάρα πολύ χαμηλό κυρίως σε θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας. Και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ε, πληρωμή των δεσμεύσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μεταφορά από άλλες γραμμές προϋπολογισμού, όπου ε, ε, δεν έχουν αφομοιωθεί τα κονδύλια και προτείνεται και από εκεί και πέρα τροποποίηση του κανονισμού. Μέχρι να εξαντληθούν τα κονδύλια βέβαια, μπορεί να ε, υπάρξουν αρκετές εβδομάδες καθυστέρηση. Ακριβώς λόγω αυτής της λύσης ε, υπήρξαν πολλέ περιπτώσεις, κυρίως σε θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας, που δεν μπόρεσαν να καταβληθούν οι πληρωμές. Ε, επειδή ακριβώ υπάρχουν πάρα πολλέ καθυστερήσει και αποπληρωμέ από προηγούμενα χρόνια, έχουμε καθυστερήσει επί των καθυστερήσεων και αυτά συσσωρεύονται κάθε χρόνο. Ε, αυτό το υψηλό ποσοστό καθυστέρηση και τη αδυναμία να καταβάλλονται τα ποσά εν ευθέτω χρόνο, κυρίω σε θέματα ανθρωπιστική βοήθεια, θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο και είναι κάτι το οποίο υποσκάπτει την ε, φήμη τη Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα τη ανάπτυξη όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου στο Συμβούλιο, σας παρακαλώ όσοι έχετε συζητήσεις να τις κάνετε εκτός αιθούσης, διότι δεν μπορούμε να ακούσουμε τον εισηγητή που μιλάει. Σας παρακαλώ τα πηγαδάκια εκτός λοιπόν, ε, διακόπτη πρόεδρος. Ευχαριστώ. Για τι διαπραγματεύσει λοιπόν Οκτωβρίου-Νοεμβρίου στο Συμβούλιο, στη διαδικασία τη συνδιαλλαγή, ο κύριο Ρούμπιχ προτείνει η Επιτροπή Ανάπτυξη να έχει μια πολύ αυστηρή θέση και να μην επιτρέψει να γίνουν περικοπέ ε, στον τομέα τη ε, ε, ανάπτυξης ε, και θα πρέπει οι δεσμεύσεις να είναι αντίστοιχες με τις πληρωμές. Και επειδή θέλουμε να έχουμε μια ισχυρότερη διαπραγματευτική θέση, ο κύριος Ρούμπιχ προτείνει να θεωρήσουμε ότι είναι προτεραιότητα αυτό για την Επιτροπή Ανάπτυξης και να επικεντρωθεί σε αυτό και ταυτόχρονα να δεχτεί κάποιες πολύ μικρές περικοπές οι οποίες προτείνονται από το Συμβούλιο ως ε, τακτική προσέγγιση. Κάποιες από τις περικοπές οι οποίες προτείνονται είναι για παράδειγμα περικοπές ε, στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας, του μέσου αναπτυξιακής συνεργασίας, αντί των 2 εκατομμυρίων που προτείνονται να δεχτούμε 1 εκατομμύριο για παράδειγμα και σε κάποια άλλα προγράμματα προτείνει αντίστοιχη προσέγγιση. Μία ακόμα προτεραιότητα την οποία θα ήθελε να επισημάνει ο κύριος Ρούμπιχ, είναι ε, το αποθεματικό εκτάκτου ανάγκης. Ε, ξέρουμε ότι οι ανθρωπιστικές κρίσεις τα τελευταία χρόνια είναι όλο ένα και πιο αυξημένες και φυσικά αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. το αποθεματικό εκτάκτου ανάγκης είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο το οποίο μπορεί να προβλέψει ε, κονδύλια για ξαφνικές και απρόβλεπτες κρίσεις και ενισχύεται αυτό. Η άποψη λοιπόν του κυρίου Ρούμπιχ είναι η Επιτροπή ανάπτυξη να δεχτεί μικρότερες περικοπές στον προπολογισμό, αλλά να πιέσει για ε, εξίσωση πληρωμών και δεσμεύσεων, καθώς επίσης και ενίσχυση του ε, αποθεματικού αυτού του εκτάκτου ανάγκης. Ευχαριστώ. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκερέρο θέλει το λόγο. Και στη συνέχεια ο κύριος Νόιζερ. Ευχαριστώ πολύ. Ο σκιώδης ε, συντάκτης ε, εκ των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών θα ήθελα να σας επισημάνω ότι σε γενικές γραμμές συμφωνώ με τη γνωμοδότηση, αλλά θα ήθελα να κάνω τρία σχόλια. Ένα εξ αυτών έχει να κάνει με το γεγονός ότι συμφωνώ ναι, με την ιδέα ότι ο βασικός μας στόχος είναι η μείωση της ένδυας και ε, η ε, ε, ενίσχυση κάποιων ε, που είναι πιο ευάλωτοι, αλλά να μην εγκαταλείψουμε και εκείνα τα τμήματα της κοινωνίας σε κάποιες χώρες τις οποίες ναι μεν το ΑΕΠ δεν είναι τόσο επιζήμιο, μπορεί να είναι λίγο υψηλότερο το ΑΕΠ, αλλά υπάρχουν κάποιες κοινότητες, κάποιες περιοχές, κάποια τμήματα της κοινωνίας λόγω φύλου, λόγω ηλικίας που βρίσκονται σε δεινότερη κατάσταση και θα πρέπει φυσικά να ληφθούν και αυτοί υπόψη στα πλαίσια της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δεύτερη ε, ανησυχία μου και θα ήθελα να συγχαρώ και τον συντάκτη της γνωμοδότησης γι' αυτό είναι ε, το θέμα της εξίσωσης μεταξύ των διαθέσιμων πόρων και των δαπανών. Διότι αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει ένα έλλειμμα και το έλλειμμα αυτό διότι το έλλειμμα στην ε, περίπτωση της ανάπτυξης ε, και συνεργασίας δεν ε, σημαίνει ότι δεν βοηθούμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Δεν φτάνουν τα χρήματα σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Γι' αυτό λοιπόν οι δεσμεύσει υποχρεώσεων και οι δεσμεύσει πληρωμών και οι υποχρεώσεις πληρωμών θα πρέπει να είναι εξίσου ε, κατανεμημένα ποσά. Δεν παρουσίασα καμία τροπολογία επί του θέματος, αλλά υπάρχει και ένα θέμα το οποίο θεωρώ ότι είναι ε, λαμβάνει πολύ υπόψη του το Συμβούλιο. Λέει ο κύριος Ρούμπιχ ότι κάποιες περικοπές που προτείνει το, το Συμβούλιο είναι αποδεκτές. Νομίζω ότι εδώ στην Επιτροπή μας το να δεχτούμε ότι στη συνεργασία για την ανάπτυξη σε αδρές γραμμές είναι δεκτές κάποιες περικοπές δεν αποτελεί καλή τακτική θεωρώ ότι ε, θα μπορούσαμε να πούμε το ίδιο πράγμα με τελείως αντίστροφο τρόπο. Δηλαδή να πούμε ότι δεχόμαστε τις περικοπές μόνο εάν γίνει το τάδε. Αλλά η γενικότερη στάση μας θα πρέπει να είναι ότι εδώ στην Επιτροπή δεν δεχόμαστε περικοπές. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νόιζερ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω ότι ο φίλος μου είπε αυτά που ήθελα να πω και εγώ. Σε γενικές γραμμές υπάρχει μια ε, συμφωνία σε σχέση με τις ε, περικοπές ε, που προτείνει το Συμβούλιο και την εξίσωση αυτών με αυξήσει σε άλλα κονδύλια. Ανάμεσα τώρα στον εισηγητή και στην δική μας ομάδα κατόρθωσαμε να συμφωνήσουμε σε ορισμένα σημεία για την αναπτυξιακή βοήθεια, δηλαδή να δεχτούμε τις περικοπές σε ορισμένα σημεία και αυτό αφορά τις ε, τροπολογίες 5544 και 5555. Εμείς ε, ως πολιτική ομάδα είμαστε κατά των περικοπών στην ανθρωπιστική βοήθεια επί της ουσίας, όμως ε, μπορούμε να συμφωνήσουμε στις συγκεκριμένες ως Επιτροπή Ανάπτυξης. αυτό που πρέπει να φροντίσουμε είναι να μην συμφωνήσουμε, να μην εγκρίνουμε περικοπές γενικότερου χαρακτήρα. Το Συμβούλιο φυσικά πρέπει να συνεδριάσει με την αρμόδια επιτροπή, την Επιτροπή Προεπολογισμού. Όμως πιστεύω πως εμείς ως Επιτροπή Ανάπτυξης δεν θα πρέπει να δεχτούμε στην ψηφοφορία ε, περικοπές οι οποίες θα περάσουν μετά στην Επιτροπή Προπολογισμού. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ Καλά, δεν νομίζω να υπάρχει κανένα άλλο σκιώδη συζητητή άλλων ομάδων που να θέλει να μιλήσει. Δεν νομίζω. Όχι. Κανεί άλλο δεν θέλει. Θέλετε να επανέλθετε. Με συγχωρείτε. Ναι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κ. Κάρλο Άιτ. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη θαυμάσια δουλειά που έκανε καθώς και τα διάφορα μέλη που κατέθεσαν ανθρωπολογίες. Πιστεύω ότι πράγματι τώρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση κρίσης και ο προτινόμενος προπολογισμό για την επόμενη χρονιά ήδη είναι ένας πολύ μειωμένος προπολογισμό που έχει δεχθεί περικοπές το να δεχθούμε επιπλέον περικοπέ τη τάξη των 200 εκατομμυρίων ε, στα πλαίσια τη Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟΣ, όπω προτείνει το Συμβούλιο, θα αυξήσει τι περικοπέ. Αυτή τη στιγμή πιστεύουμε ότι θα τελειώσει η χρονιά με 1,2 δισεκατομμύρια έλλειμμα. Εάν λοιπόν περάσει το ΠΕΡΕΣ 3, τότε θα περάσουμε στο 1 δισεκατομμύριο. Αλλά το γεγονός παραμένει ότι εκτιμάται ότι θα έχουμε έλλειμμα του προπολογισμού 1,2 δις. Οι περικοπές του Συμβουλίου των 200 εκατομμυρίων θα αυξήσουν αυτόν τον αριθμό. Και κανονικά, αν τα πράγματα δεν αλλάξουν, ε, θα ξεκινήσει η χρονιά ήδη με το μισό προπολογισμό. Αυτό θα έχει τεράστιε συνέπειες για τις πολιτικές που θέλουμε να εφαρμόσουμε. Θα έχει τεράστιε συνέπειες για τους διαφόρους εταίρου μας, είτε είναι ΜΚΟ, είτε διεθνεί οργανισμοί, είτε εταιρείε. Και το πιο σημαντικό και σοβαρό είναι ότι τα άτομα που θέλουμε να βοηθήσουμε, εκείνα θα θυγούν. Και αυτό θα έχει και πολιτικές συνέπειες, εφόσον σε ορισμένες χώρες όπου δεν μπορούν να καλυφθούν αυτά τα κενά του προπολισμού, θα βγουν εκτός τροχιάς ε, και δεν θα μπορούν να ακολουθήσουν τις πολιτικές τους. Σας ευχαριστώ λοιπόν για όλες τις τροπολογίες που έχουν σαν αντικείμενο να αποκατασταθεί η κατάσταση. Αναφορικά τώρα με τις πιστώσεις δεσμεύσεων. Νομίζω ότι εμείς μπορούμε να δεχθούμε τις μικροπερικοπές που προτείνονται έτσι κι αλλιώς. Εάν συνεχίσουμε έτσι, με το να θέλουμε πάση θυσία να εκτελέσουμε το μέγιστο προπολογισμό χωρίς να διαθέτουμε τα μέσα για να καταβάλουμε τις πληρωμές και να ελοπίσουμε τις πολιτικές, Βαίνουμε προς την καταστροφή. Γι' αυτό συνιστώ σύνεση σήμερα το πρωί στην Επιτροπή του Προπολογισμού, φαντάζομαι ότι ελέγχθηκε αυτό, δεν πρέπει να συνεχίζουμε να θέλουμε από τη μια πλευρά να συνεχίσουμε την πολιτική που είχαμε πάντοτε και από την άλλη πλευρά να μην έχουμε τα μέσα για να υλοποιήσουμε αυτή την πολιτική. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θέλετε να επανέλθετε. Θα είμαι πολύ σύντομα, κυρία Πρόεδρε. Απλώς, για να υπογραμμίσω, μετά από τη συζήτηση είδαμε ότι μπορούμε να καταλήξουμε ότι έχουμε τον ίδιο στόχο. Ίσως οι τακτικές του κυρίου Ρούμπικη είναι λίγο διαφορετικές. Αλλά θα μπορούσαμε, εκεί ίσως δεν συμφωνούμε ίσως με τις τακτικές, αλλά λόγω του γεγονότος, όπως ξέρουμε πολύ καλά προς τα που πηγαίνει το Συμβουλίο, η τακτική που προτείνει είναι ρεαλιστική και υπογραμμίζω για μία ακόμη φορά ότι η Επιτροπή αυτή δεν θα πρέπει να επιτρέψει ε, περικοπές ε, στις πληρωμές ε, για να αντισταθμίζουν τις δεσμεύσεις. Τελικά ε, αυτό είναι ο σκοπός μας και νομίζω ότι αυτό πρότεινε ο κύριος Ρούμπικ και τον υποστηρίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών είναι αύριο μέχρι τις 6 ώρα όσον αφορά αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης και η ψηφοφορία θα γίνει στις 23 Σεπτεμβρίου. Ευχαριστώ πολύ. Ας περάσουμε τώρα στην ψηφοφορία της Νέας Επιτροπής. Έχετε τις ε, καρτέλες σας δεν θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά παρά μόνο αν χρειάζεται παλήθευση. Θα κάνουμε μια δοκιμή για να δούμε αν λειτουργούν τα μηχανήματα. Κάντε ό,τι θέλετε, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί για να δείτε αν λειτουργεί το σύστημα. Κοιτάξτε αν λειτουργεί το σύστημά σας. Εντάξει, αρχίζει η ψηφοφορία. Λειτουργούν τα μηχανήματά σας. Τα ελέγξατε. Κλείνει η ψηφοφορία τώρα. Λειτουργούν τα μηχανήματά σας. Όλοι ψήφισαν πολύ καλά. Προχωράμε λοιπόν. Αρχίζει η ψηφοφορία. θα ακολουθήσουμε τη λίστα. Πρώτα έχουμε διορθώσεις από τον κύριο Γκερέρο, ο οποίος επιθυμεί να κάνει μια διόρθωση. Εάν δείτε το κείμενο που έχετε μπροστά σας, θέλει να αλλάξει αυτό που λέει υπό ε, τα προγράμματα των χωρών που καλύπτουν και να πει υπό το DCI που θα αφορά τις βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, εστιάζοντας ε, στην υγεία και την παιδεία και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτό δεν υπάρχει στον κατάλογο, αλλά ελπίζω να το καταλάβατε. Είδατε ποια είναι η προτινόμενη διόρθωση, εντάξει. Πολύ καλά. Ας ψηφίσουμε λοιπόν το 210201. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτό. Δεκτή. Ήταν η 55 5500 η τροπολογία. Λοιπόν, η επόμενη. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 55 Πηγαι5-10 του κύριου Νόιζερ Ποιοι είναι υπέρ. Όχι, όχι, είναι το. All those against. Ποιοι είναι κατά. Θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. vote is open, sorry. The vote is closed. Κλείνει η ψηφοφορία. έγινε, πέρασε η τροπολογία 15 με 10. Ε, αργούμε λίγο επειδή είναι η πρώτη διαδικασία ηλεκτρονική και παίρνει λίγο χρόνο που να συνηθίσετε. Ακόμα και για μένα είναι η αρχή. Λοιπόν, ας έρθουμε τώρα στο 5542. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 5542. Κατά. Θα το επαληθεύσουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. The vote is closed. Κλείνει. Ναι, δεκτή. 15 προς 11. Προτείνεται οι, οι επόμενες από το 5511 μέχρι την 5519 να ψηφιστούν συνολικά. Ε, αν δεν έχετε αντίρρηση, ψηφίζουμε συνολικά. Συμφωνείτε? Πολύ καλά. Λοιπόν, ποιοι είναι υπέρ αυτού του συνόλου των τροπολογιών. Κατά. Αποχές. Δεκτές. Ευχαριστώ πολύ. Amendment 5. Τροπολογία 5543 του κυρίου Νόιζερ. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσαμε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται 13 ψηφιπέρ, 12 κατά. Επόμενη, 55-20. Καταπίπτει. 55-21. Ποιος είναι υπέρ. «55-21 και 55-01 μαζί. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 55-22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μία άλλη πρόταση για να ψηφίσουμε σε μπλοκ από την 55.23 μέχρι την 55 από τους Noiser Gerents Venter. Συμφωνείτε όλοι να ψηφίσουμε σε μπλοκ. Ωραία. Ποιοι είναι υπέρ της ψηφοφορίας σε μπλοκ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5504 της κυρίας Σλάιν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5505 της κυρίας Σλάιν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 55-48 του κυρίου Μισελ. Υπέρ. Κατά. Δια... Αποχές. Εγκρίνεται. 55-50 του κυρίου Νόιζερ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 55-52 από τους κύριους Ρούμπι και Βέντα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άλλη μια πρόταση για ψηφοφορία σε μπλοκ από την 5506 μέχρι την 5507. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, αποχές, εγκρίνεται. 5540 του κύριου Νόιζερ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται με 15 ψήφους υπέρ, 12 κατά. Η 5508 καταπίπτει, 5531 άρχεται η ψηφοφορία. Με συγχωρείτε λέει πρόεδρος, ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Και εγώ πρώτη φορά κάνω ψηφοφορία. 55-32. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 55-49 του κυρίου Νόιζερ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άλλη μια ψηφοφορία σε μπλοκ από την 55-33 μέχρι την 55-35. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά αποχές εγκρίνονται. 55-44 του κυρίου Νόιζερ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Η ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ίδια πλειοψηφία 15 προς 12 εγκρίνεται. 55-45 υπέρ, κατά, θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνατε πάλι με 15 ψήφους υπέρ, 12 κατά. Επόμενο μπλοκ από 55-36 μέχρι 55-38. Το δέχεστε όλοι. Ποιοι είστε υπέρ. Ποιοι κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Τελική ψηφοφορία από τους κυρίους Νόιζερ και Γκέρενς. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή κύριο Ρούμπε και όλους ε, τους και οδησηγητές και όσοι εργάστηκαν για την ψηφοφορία αυτή. Τώρα, Κερδίσαμε χρόνο, αγαπητοί συνάδελφοι, και πρέπει να περιμένουμε την ε, Επίτροπο. Α, μάλιστα, είναι ήδη εδώ, υπέροχα. Παρακαλώ καθίστε τότε και θα καλωσορίσουμε την Επίτροπο. Okay, can I ask everyone to take... Λοιπόν, καθίστε παρακαλώ. Σας παρακαλώ, όσοι είναι όρθιοι και συζητούν, παρακαλώ καθίστε ή περάστε έξω να συνεχίσετε τις συζητήσεις σας. Παρακαλώ, συναδελφοί, καθίστε ή περάστε έξω για τις συζητήσεις σας. Το αυτό ισχύει και για όσους βρίσκονται στο πίσω μέρος της αίθουσας. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε την τιμή λοιπόν να καλωσορίζουμε εδώ την Επίτροπο Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, η οποία είναι Επίτροπος Αρμόδια για την Ανθρωπιστική Βοήθεια στη συνεδρίασή μα. Είναι η δεύτερη συνεδρίαση τη Επιτροπή μα εδώ στο Κοινοβούλιο. Έχουμε ε, ξανασυναντηθεί. Ήρθατε και πριν από τι καλοκαίρινέ διακοπέ και χαιρόμαστε που μπορείτε να έρθετε τόσο σύντομα και πάλι ήσασταν ιδιαίτερα δραστήρια με το Κοινοβούλιο και στην προηγούμενη θητεία, γνωρίζω ε, από τους συναδέλφους και δείξατε αμέσως ότι είστε διαθέσιμοι και ξέρω ότι πιέζεστε ιδιαίτερα. Μιλήσαμε και σήμερα το πρωί ε, για το θέμα αυτό, παρά το γεγονός ότι κάποιοι από εμά είχαμε καλές καλοκαιρινές διακοπές, για πολλούς άλλους ανθρώπους ε, σε όλο τον πλανήτη δεν ήταν τόσο ευχάριστο το καλοκαίρι. Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τόσο μεγάλη ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας ε, και δεν ήταν τόσο δραστήρια η ΕΚΟ. Ξέρω, κυρία Επίτροπε, ότι και εσείς ήσασταν ιδιαίτερα δραστήρια στη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών. Ε, είχαμε δει και το Γενικό Διευθυντή σας, τον Κλάς Σόρενσεν, ο οποίος μας μίλησε για το μέλλον της ανθρωπιστικής βοήθεια και τους στόχους που μας περιμένουν. Νομίζω ότι ούτε τότε δεν είχαμε αντιληφθεί πόσο σοβαρές ήταν αυτές οι προκλήσεις και σήμερα το πρωί έγινε μια συζήτηση για τη Γάζα Ψηφίσαμε μόλις και τον προϋπολογισμό για το επόμενο έτος και αντιλαμβανόμαστε πολύ ε, καλά τα σοβαρά προβλήματα στον προϋπολογισμό που αντιμετωπίζει το δικό σα το τμήμα και θα μας μιλήσετε φαντάζομαι και γι' αυτά. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε τις απόψεις σας και να δούμε αν ε, μπορεί να σας βοηθήσει με τον οποιονδήποτε τρόπο η Επιτροπή μας, ώστε να φτάσει ανθρωπιστική βοήθεια σε όλους. Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Για όσους επανεξελέγησαν ή εξελέγησαν για πρώτη φορά, συγχαρητήρια. Η Επιτροπή σας είναι μία από τις επιτροπές η οποία θα έχει όλο και περισσότερη σημασία για την θέση της Ευρώπης ανά τον κόσμο, αλλά και για την προστασία των ίδιων μας των πολιτών, διότι οι κρίσεις ε, στις οποίες αναφερθήκατε ε, σε μεγάλο βαθμό αφορούν και ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στην εγγύης γειτονία, αλλά και ανθρώπους οι οποίοι ε, φτάνουν και στην Ευρώπη. Και ξέρουμε ότι φτάνουν ε, στο κατόφλι μας, αλλά πολλές φορές όχι με λουλούδια, αλλά ε, δυστυχώς κομίζουν άσχημα νέα. Θα ήθελα λοιπόν εν συντομία να σας πω πώς βλέπω εγώ το χαρτοφυλάκιο αυτό, διότι είμαι και μια επίτροπος η οποία φεύγει εντός ολίγου, γιατί κάνουμε τι και τι στάση τηρούμε στις βασικές κρίσεις και να πούμε και δύο λόγια στο πλαίσιο αυτό, τα οποία θεωρώ ότι θα είναι σημαντικά για το έργο της Επιτροπής σας. Θα ήθελα να ξεκινήσω λοιπόν με την πρώτη ε, παρατήρηση, η ανθρωπιστική βοήθεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η ανθρωπιστική βοήθεια πιο συγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως γνωρίζετε ήδη από το Γενικό Διευθυντή μας, ε, είναι η πρώτη φορά που η Ευρώπη έχει ε, έναν επίτροπο αρμόδιο για την ανθρωπιστική βοήθεια και επίσης είναι και η πρώτη φορά που συνενώνουμε δύο μέσα, το Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και την Ανθρωπιστική Βοήθεια. Εκ έχω διαπιστώσει ότι είναι πολύ ε, σωστή αυτή η απόφαση, διότι βρισκόμαστε σε έναν κόσμο ο οποίος πλήττεται από όλα και πιο καταστροφικές ε, και θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο πώς μπορούμε να δράσουμε σε κατεπίγουσε περιπτώσεις, αλλά και πώς μπορούμε το μέσο της ανθρωπιστικής βοήθειας να το χρησιμοποιήσουμε και ή δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε και τις εγγενείς δυνατότητες ε, ε, σε είδος των κρατών μελών μας. Και θα σας δώσω και αυτά παραδείγματα του πώς εφαρμόζονται αυτά. Ο βασικός μας στόχος είναι να δώσουμε βοήθεια σε θύματα καταστροφών και ε, θύματα ενόπλων σειράξεων ε, όλα ε, επί τη βάση της ανθρωπιάς, ε, της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας. Και νομίζω ότι ο κόσμος χρειάζεται περισσότερο και όχι λιγότερο σεβασμό για αυτές τις αρχές. Έχουμε να διαδραματίσουμε ένα ρόλο ο οποίος είναι τρισδιάστατος. Πολιτική, επιχειρήσεις και προάσπιση των όσων κάνουμε. Αυτό το οποίο προβάλλεται περισσότερο φυσικά είναι οι επιχειρήσεις μας. Αλλά οι πολιτικές μας έχουν σημασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν στην πρώτη γραμμή εφαρμογής συγκεκριμένων πολιτικών στην ανθρωπιστική βοήθεια, οι οποίες εφαρμόστηκαν ε, φαγμιδών, όπως για παράδειγμα επισητιστική βοήθεια, σε είδος, δηλαδή ε, δίνοντας τα γεωργικά μας πλεονόσματα σε χώρες ε, και σε μετρητά, δηλαδή βοηθήσαμε και τις τοπικές κοινωνίες αλλά και τους γεωργούς και τις τοπικές αγορές ώστε να μπορούν να βοηθήσουν τους εαυτούς τους και να μην βασίζονται στη βοήθεια κάθε χρόνο η πολιτική η οποία θεωρώ ότι ήταν ιδιαίτερα σημαντική και για σήμερα αλλά και για το μέλλον είναι η πολιτική μας για την αποφασιστικότητά μας, ε, δηλαδή να βοηθήσουμε ε, κοινότητες σε διάφορες χώρες για να μπορέσουν να αντέξουν τα διάφορα σοκ, να μειώσουμε τον αριθμό των σειράξεων, να μειώσουμε τους κινδύνους από τις φυσικές καταστροφές, ε, για να μην εξαφανιστούν χρόνια αναπτυξιακής πρόοδου και ελπίζω ότι αυτά θα είναι περισσότερο και όχι λιγότερο σημαντικά στο εγγύς μέλλον. Από επιχειρησιακή σκοπιά ε, δίνουμε περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ σε ετήσια βάση ανθρωπιστικής βοήθειας σε περίπου 200 ε, ανθρωπιστικές οργανώσεις, εταίρους μας. Και αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να τονίσουμε ότι σύντο χρόνο έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε ένα σταθερό δίκτυο Όλο και περισσότεροι άνθρωποι από την ομάδα μου βρίσκονται στα σημεία στα οποία έχουμε θερμά επεισόδια στη πλανήτη και όχι στις Βρυξέλλες. Έχουμε 250 άτομα στα 44 επιτέπου γραφεία που μπορείτε να δείτε στο χάρτη. Και αυτό το οποίο θα διαπιστώσετε, είμαι βέβαιη, είναι ότι η συγκέντρωση αυτών των επιτόπιων γραφείων είναι όντως εκεί που χρειαζόμαστε περισσότερο ανθρωπιστική βοήθεια και είναι πιο σοβαρές οι ανθρωπιστικές ανάγκες. Το δίκτυο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μα. είναι πολύτιμο για να μπορέσουμε να δώσουμε προτεραιότητε και να διοχετεύσουμε καταλήλω του πόρου μα, και είναι εξίσου σημαντικό και για του φορολογουμένους, διότι αυτοί οι άνθρωποι είναι τα μάτια και τα αυτιά των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Επικεντρωνόμαστε στην αποτελεσματικότητα, στην αποτελεσματική χρήση πόρων και κάθε χρόνο ελέγχουμε το 1 τρίτο των προγραμμάτων μας και το 1 τρίτο των εταίρων μας, ώστε να είμαστε ε, βέβαιοι ότι υπάρχουν αποτελέσματα για τη βοήθεια που παρέχουμε. Είμαστε μια σπάνια περίπτωση υπηρεσίας που έχει εξετάσει πάρα πολύ προσεκτικά πώς λειτουργεί. Έγινε και μία αναθεώρηση ε, ως προς τη λειτουργία μας ε, και είχαμε 20% περίπου βελτίωση στην αποδοτικότητά μας ε, εξαιρώντας ε, διάφορες διαδικασίες που θεωρούμε ότι δεν προσδίδουν καμία αξία και εξορθολογίζοντας τον τρόπο με τον οποίο παρέχουμε ανθρωπιστική βοήθεια. Το αποτέλεσμα είναι ότι 120 εκατομμύρια και άνθρωποι κάθε χρόνο λαμβάνουν ε, συνδρομή, η οποία ορισμένες φορές τους σώζει και, για τη ζωή, και τη ζωή χάρη σε αυτά που κάνουμε με λιγότερο από το 1% του συνολικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήμασταν ιδιαίτερα δραστήριοι και έχουμε προωθήσει ε, το γεγονός ότι πρέπει να επικεντρωνόμαστε στις ανάγκες των παιδιών. Παίρνουμε τα χρήματα και δημιουργήσαμε το EU Children of Peace που είναι ένας τρόπος ε, για να ε, επικεντρώσουμε την προσοχή μας στα παιδιά γιατί δεν θέλουμε να χρησιμοποιούνται ε, οι κατεπίγουσες περιπτώσεις για να εκριζώνονται αυτά τα παιδιά από τις πατρίδες τους. Επίσης θεωρώ ότι υπάρχει υποστήριξη για τους ανθρώπους μας, ακριβώς γιατί γίνεται πολύ σκληρή δουλειά ε, από τις ομάδες αυτές. 9 στους 10 Ευρωπαίους λένε ότι υποστηρίζουν την ανθρωπιστική βοήθεια και θεωρώ ότι αυτό είναι γιατί είναι μεν δεοντολογικά σωστή η ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά γιατί ταυτόχρονα αντιλαμβάνονται ότι έχει και αξία για την προσωπική μας ασφάλεια. Θα ήθελα να ξεκινήσω από το γεγονός ότι δυστυχώς οι ανάγκες μας αυξάνονται ε, σε έναν κόσμο όπου οι πόροι μας είναι κορεσμένοι. Δεν είναι υπερβολή να σας πω ότι από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και μετά αυτή είναι η μεγαλύτερη κρίση που έχουμε διαπιστώσει και υπάρχουν και στοιχεία τα οποία ε, το επιβεβαιώνουν αυτό. Έχουμε πάνω από 50 εκατομμύρια εκτοπισμένους ανθρώπους, είτε εσωτερικός είτε πρόσφυγες και αυτό είναι μακράν ο μεγαλύτερος αριθμός που έχουμε διαπιστώσει από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τούδε αλλά επίσης κάτι το οποίο είναι εκπληκτικό, ο αριθμός αυτός αυξάνεται κάθε χρόνο και μάλιστα ε, εκθετικά. Από πέρσι ε, μέχρι φέτος είχαμε επιπλέον 6, άτομ, 6 εκατομμύρια εκτοπισμένους ανθρώπους. Είναι σαν ε, να εκτοπιστεί η μισή Ιρλανδία σε ένα χρόνο. σήμερα έχουμε τέσσερις κατεπίγουσε περιπτώσεις πέδου 3. Ο αριθμός 3 είναι ο υψηλότερο αριθμός ε, που ε, δίνεται από τον ΟΗΕ. Ε, Συρία, Ιράκ και Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία τη κεντρική Αφρικής. αυτό είναι κάτι εξαιρετικό. Συνήθω έχουμε μία τέτοια κρίση ή και δύο, αλλά ποτέ μέχρι τώρα δεν είχαμε τόσο ε, μεγάλες κρίσεις. Και όπως βλέπετε δεν αναφέρω εδώ ούτε την Ουκρανία, ούτε τη Γάζα, ούτε τον Εμπόλα, ούτε τη Σομαλία που έρχεται και αυτή στο προσκήνιο. Ε, υπάρχουν κρίσεις λοιπόν οι οποίες είναι πάρα πολύ οξύες. Και αυτό το οποίο θα πρέπει να αναγνωρίσουμε είναι ότι η κρίση μάλλον οι κρίσει είναι αλληλένδετε. Ανηφερόμαστε στην κάθε μία ξεχωριστά, αλλά φαίνεται ότι σιγά σιγά υπάρχει σχέση μεταξύ των. Και δυστυχώς ε, η αστάθεια, η αλλαγή του ε, κλίματος και ο εξτρεμισμό δεν ε, καθιζάνουν. Είναι κάτι το οποίο δημιουργούν ολοένα και περισσότερες ανάγκες. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω με το πρώτο κύμα κρίσης ε, σε αυτό το κατεπήγον ε, ποσοστό 4. Βλέπετε ότι εδώ έχουμε τη Συρία και το Ιράκ. Η κρίση της Συρίας εξακολουθεί να βαθαίνει. Έχει πέσει από το, η ιεραρχία στις προτεραιότητές μας, αλλά το τελευταίο διάστημα ήταν από τις πιο καταστροπτικές και από πλευράς βίας και από πλευράς ε, απώλειας ανθρωπίνων ζωών από τότε που ξεκίνησε η κρίση. 10,8 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται πλέον βοήθεια και πριν από λίγες μέρες δυστυχώς περάσαμε το ε, λυπηρό όριο των 3 εκατομμυρίων προσφύγων σε γειτονικές χώρες. Από την αρχή της κρίσης αυτής η Ευρωπαϊκή Ένωση βρισκόταν στην πρώτη γραμμή. Είμαστε ο μεγαλύτερος δωρητής ανθρωπιστικής βοήθειας. Έχουμε δώσει μέχρι τώρα 2,8 δις ευρώ και συνεχίζουμε να κάνουμε δύο πράγματα. Να συγκεντρώνουμε πόρους για τους ανθρώπους εντός της Συρίας, για τους πρόσφυγες αλλά και για τις ε, ε κοινότητες τις τοπικές και ταυτόχρονα πιέζουμε και τους υπολείπους να κάνουν περισσότερα. Στις 23 Σεπτεμβρίου θα συμπροεδρεύσω σε μια συνεδρίαση για τη Συρία ε, με ε, στόχο να έχουμε δωρητές και χορηγούς και ε, κυρίως ζητάμε από άλλες χώρες να κάνουν περισσότερα. Επίσης έχουμε επιμείνει πολύ σε αυτή την κρίση και σε άλλες για το συντονισμό και την αποτελεσματική απάντησή μας στα διάφορα θέματα. Αυτό το θέμα του συντονισμού όσες φορές και να το επαναλάβουμε δεν αρκεί γιατί ο μεγάλος κίνδυνος που ελοχεύει σε περίπτωση κρίσεων είναι να ε, ε, βοηθήσουμε κάποιους ανθρώπους δύο και τρεις φορές και κάποιους άλλους καθόλου. Και φυσικά αυτός ο συντονισμός ε, πρέπει να είναι βιώσιμος και της βοήθειας των τοπικών κοινοτήτων και εκεί μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερα πέραν των χρημάτων μας. Για τη Συρία ανησυχούσαμε ευθύ εξ αρχή και κάποια μέλη τη Επιτροπή ε, θυμούνται κάποιε συζητήσει επί του ζητήματο ε, ε, και ξέραμε ότι θα υπάρχει και διάχυση του φαινομένου και αυτό το οποίο μα ανησυχούσε περισσότερο είναι να υπάρξει κάποιο αντίστοιχο φαινόμενο στο Λίβανο ή και στην Ιορδανία κάποια αποσταθεροποίηση. Αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ Συρίας και Ιράκ και μάλιστα με πολύ δραματικό και επικίνδυνο τρόπο. Στο Ιράκ ε, μετέβην το Μάρτιο και είδα ε, το, ε, το πόλεμο μεταξύ Σουνιτών Σιητών. Έκτοτε υπήρχε και μια διάχυση από τη Συρία στο Ιράκ ε, εδώ έχουμε τον Ισλαμικό, το Ισλαμικό κράτος και εδώ έχουμε την πιο βάναυση και πιο ε, καταστρεπτική μηχανή θανάτου που υπάρχει αυτή τη στιγμή ε, στον κόσμο. Δράσαμε πολύ γρήγορα. Ήδη από το Μάρτιο αποφασίσαμε να ανοίξουμε γραφείο εκεί, μια υπηρεσία δίνουμε πολλά χρήματα, αλλά ταυτόχρονα χρησιμοποιείται και το μέσο της πολιτικής προστασίας, διότι οι εκτοπισμένοι στο Ιράκ ε, εκτοπίστηκαν με τόσο γρήγορο τρόπο, ώστε το να ε, γίνουν τα χρήματα αγαθά και βοήθεια δεν αρκεί. ενεργοποίησαμε την πολιτική προστασία, ζητούμε δηλαδή ε, στήριξη σε είδος από τα κράτη-μέλη και έχουμε ήδη 20 ε, ανθρωπιστικές πτήσεις ε, που έχουν στείλει πολλά βοήθεια. Καταφέραμε λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο για να δώσει ταχύτατα βοήθεια. Και φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να επισημάνουμε ότι τα τελευταία δύο χρόνια προσπαθούμε να πείσουμε ε, οι νέοι δωρητές του κόλπου να είναι πιο δραστήριοι για να μπορέσουν να δώσουν περισσότερα και καταφέραμε το βασίλειο της Σαουδικής ε, Αραβίας να δώσει 500 εκατομμύρια δολάρια για πρώτη φορά μέσω του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και καλό θα ήταν να ακολουθήσουν και άλλοι το παράδειγμά τους, αλλά πραγματικά εκεί ε, μας προσφέρεται και μια μεγάλη ανακούφιση. Και βέβαια πρέπει να είμαι ειλικρινής και να σας πω ότι παρά τη βοήθεια που παρέχουμε, στην καλύτερη δεύτερη περίπτωση βοηθούμε ανθρώπους που βρίσκονται στο κουρδικό τμήμα και σε περιοχές στις οποίες έχουμε πρόσβαση στο νότιο Ιράκ. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο τμήμα γης ε, στο Ιράκ το οποίο ε, είναι εντελώς ε, απροσπέλαστο και εκεί το Ισλαμικό κράτος έχει τα ενία και κατά την άποψή μας 500.000 άνθρωποι περίπου είναι άνθρωποι στους οποίους δεν έχουμε καμία πρόσβαση. Τι θα συμβεί τώρα στις επόμενες εβδομάδες και μήνες ε, θα δούμε, αλλά σίγουρα ελοχεύει πάρα πολύ σοβαρός κίνδυνος ε, για τον ε, αυτόχθονο πληθυσμό, κυρίως για μειονότητες και μειονότητες οι οποίες δεν βρίσκονται μεν επιτόπου, αλλά είναι επικίνδυνες. Να περάσω τώρα σε μια άλλη ζώνη κρίσης. Ναι. Πρόκειται για το, την κεντροαφρικανή δημοκρατία και το Νότιο Σουδάν, επίπεδα 2 και 3 επίγουσα κατάσταση. Πρωτού μιλήσουμε για την Αφρικανική Δημοκρατία. Κοιτάξτε αυτή τη λωρίδα που ξεκινάει από το Μαλί, πηγαίνει στην Βόρειο Νιγηρία, περνάει από το Καμερούν, πηγαίνει στη Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, στο Νότιο Σουδάν, Σομαλία και βεβαίω βλέπετε πού καταλήγει. Και εδώ δεν περιλαμβάνουν τη Λιβύη, διότι περιοριζόμαστε σε αυτά όσα κάνουμε από πλευρά ανθρωπιστική βοήθεια στη Λιβύη. Αυτές οι δύο γειτονικέ χώρες, η, το Νότιο Σουδάν και η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, αντιμετωπίζουν φοβερέ καταστάσεις και ο φόβος μου είναι ότι επειδή η προσοχή στρέφεται όλο και περισσότερο προ το Ιράκ, δεν υπάρχει αρκετή προσοχή σε αυτή την περιοχή. Και όμω το Νότιο Σουδάν υπάρχει μεγάλη ανθρωπιστική καταστροφή. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται ε, σε απελπιστική κατάσταση επειδή αυτοί που βρίσκονται στην εξουσία είναι κατάλληλοι και ελπίζουμε ότι θα αποφευχθεί ένας λοιμός. Ελπίζουμε να μην υπάρξει λοιμός. Και πέραν από ε, την προσοχή μας που είναι στραμμένη προς τα εκεί και τη βοήθεια που παρέχουμε, πιστεύουμε ειλικρινά ότι αυτή είναι ακόμη μια περίπτωση όπου είναι η ευθύνη και της κυβέρνησης και των ανταρτών να φροντίσουν ε, τα άτομα τα οποία έχουν αμελήσει στην Κέντρο Αφρικανική Δημοκρατία. Εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση από την πρώτη μέρα είχε δραστηριοποιηθεί από τη στιγμή που άρχισαν τα προβλήματα και να ταραχές όταν ξεκίνησε αυτή η σύγκρουση μεταξύ των θρησκειών στρέψαμε την προσοχή μας προς τα εκεί και αναλάβαμε δεσμεύσει σε εμείς Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της ασφάλειας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ταμείο ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με τη συμμετοχή των κρατών μελών με την ελπίδα να χρησιμοποιήσουμε με ένα νέο τρόπο τους πόρους μας προκειμένου να ε, είναι ο, ο τρόπος να χρησιμοποιηθούν συντονισμένος. Το πρόβλημα της ασφάλειας είναι πολύ σημαντικό, όχι μόνο για να βγει η χώρα από αυτή την κατάσταση, αλλά γενικά η ασφάλεια είναι απαραίτητη. Και βλέπετε τα δύο κόκκινα σημεία στο χάρτη. Τα επισημένο είναι τα πιο ορατά και παρόλο ότι δεν είναι οι μόνες ε, θερμές περιοχές στην Αφρική. Ας περάσω τώρα στον, ε, στην επιδημία του έμπολα. Είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί όλους, σε όλες τις χώρες. Γνωρίζετε τα γεγονότα, τι έχει συμβεί. Ε, υπάρχουν τόσοι νεκροί και πόσες χώρες έχουν πληγεί. Πέντε χώρες τώρα που έχουν ε, ε, περιπτώσεις, περιστατικά στην επικράτειά τους. Και είναι η Λιβύη, η Σιεραλεόνη και η Σενεγάλη. Γιατί είναι διαφορετική έμπολα από άλλες πανδημίες. Είναι η πρώτη φορά που υπάρχει πανδημία σε χώρες που δεν έχουν συστήματα υγείας για να την αντιμετωπίσουν οι χώρες που μόλις έχουν βγει από συγκρούσεις, ε, χώρες που χαρακτηρίζονται από αστάθεια και όλες οι αντιδράσεις είναι εξωστρεφείς, εξωγενείς. Ε, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας προσπαθεί να βοηθήσει και εμείς δώσαμε 11,9 εκατομμύρια ευρώ και μας λένε «Μα αυτά δεν αρκούν. Μα το σημαντικό είναι ότι αυτά τα χρήματα έχουν δοθεί για αυτό το σκοπό, για να σταματήσει στην πηγή το κακό. Αυτή τη στιγμή έχουν σταλεί εμπειρογνώμονές μας στις ε, τρεις χώρες, ε, Γουινέα, Σιεραλιώνη και Λιβύη, για να μπορέσουμε να παράσχουμε ανθρωπιστική βοήθεια και για να αποχωρήσουν οι άρρωστοι. Επίσης, θα ζητήσω να δοθούν ε, και παγκοσμίω και από την Αμερική χρήματα. 200.000 έχουν δοθεί από την Παγκόσμια Τράπεζα και 240.000 από το EDF και θα ζητήσουμε και στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο να σταλούν αυτά τα χρήματα υπό μορφή ανθρωπιστικής βοήθειας και μόνον. Το Εκείνο που είναι γνωστό είναι ότι όταν υπάρχουν τέτοιες ε, ευαίσθητες καταστάσεις, ε, είναι πρόσφορο έδαφος για να δημιουργηθούν τραγωδίες. Θα ήθελα να ολοκληρώσω με την Ουκρανία. Να μην μιλήσουμε για τη Γάζα. Η Ουκρανία τώρα. Οι εξελίξεις είναι πολύ ανησυχητικές. Από την πρώτη μέρα όταν υπήρξε αιματοχυσία στο Κίεβο, στείλαμε μια ομάδα θερπιστικής βοήθειας και από τότε βοηθάμε ε, τον Ερυθρό Σταυρό της Ουκρανίας και τώρα τις Ουκρανικές Αρχές. Ε, στείλαμε 2,5 εκατομμύρια ευρώ κυρίως για να βοηθήσουμε Ε, τη στέγαση των εκτοπισμένων. Οι αριθμοί είναι πολύ υψηλοί. Μιλάμε για τουλάχιστον 500.000 άτομα τα οποία έχουν εκτοπιστεί εσωτερικά ή προς τη Ρωσία. Αλλά το πιο ανησυχητικό στην Ουκρανία, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, είναι η πολιτικοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ήταν ατυχές το γεγονός ότι οι Ρώσοι έστειλαν αυτή την αποστολή και για να βοηθήσουν την πομπή αν θέλετε, να βοηθήσουν τους ανθρώπους και η προστασία των πολιτών κατά τη γνώμη μας είναι μείζον πρόβλημα. Μέχρι τώρα λοιπόν τι κάναμε. δεν τονίζουμε την ανθρωπιστική βοήθεια που στείλαμε εν μέρη, επειδή οι Ουκρανικές αρχές δεν θέλουν να πέσουν σε μια παγίδα εφόσον λένε οι Ρώσοι τους βοηθούν και εν μέρη επειδή πιστεύουμε υπήρχε κάποιος κίνδυνος χειραγώγησης κατά κάποιον τρόπο της ανθρωπιστικής μας βοήθειας για πολιτικούς λόγους. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ε, σωστή ηγεσία ε, από τον ε, αντιπρόεδρο Γκρόσμαν και διοχετεύει σωστά τη βοήθειά μας και ζητούν οι Ουκρανοί να δημιουργήσουν τις ικανότητες που απαιτούνται για να αντιμετωπίσουν μόνοι τα προβλήματά τους. Θα δώσουμε και άλλα χρήματα. Ήδη κοιτάμε πώς να χρησιμοποιήσουμε χρήματα από το Ταμείο Ανάπτυξης για να αντιμετωπιστούν αυτές οι αυξανόμενες ανάγκες. Τι υπάρχει κοινό σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Η ανεξιθρησκεία, η αδιαλαξία, ο μη σεβασμός ε, του, ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά και επίσης σημαντικό, η ανθρωπιστική βοήθεια είναι ε, σαν μια γάζα σε μια, πηγή, σε μια πληγή. Δεν αποτρέπει το να πληγώνονται οι άνθρωποι και δεν θεραπεύει. Ποια θα ήταν η θεραπεία, μια πολιτική λύση, μεγαλύτερη ανεκτικότητα, η δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα εξασφαλίζει μια σωστή ανάπτυξη και θα περιορίζει, όχι θα εξοδετερώνει, θα περιορίζει τις ανθρωπιστικές ανάγκες. Και εδώ, αν θέλετε, για να τελειώσω με αυτό, με τρεις παρατηρήσεις, εδώ νομίζω πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας. Πρώτα απ' όλα, να αναγνωρίσουμε ότι ζούμε σε ένα πιο ευαίσθητο κόσμο, ότι θα υπάρχουν όλο και περισσότερες ανθρωπιστικές ανάγκες και θα πετούν κινητοποίηση πόρων. Εμείς λοιπόν πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Επίσης πρέπει να ενεργούμε με περισσότερη αποτελεσματικότητα, να είμαστε περισσότερο εστιασμένοι στα αποτελέσματα. Δεύτερον, πρέπει να σκεφτόμαστε ποια είναι τα βαθιά αίτια αυτών των προβλημάτων. Είναι ότι δεν υπάρχει ένα σωστό διεθνές σύστημα διακυβέρνησης που δεν ανταποκρίνεται σε ανάγκες της εποχής μας. Πρέπει να έχουμε την ικανότητα να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε αυτές τις ικανότητες τι έχουμε σήμερα λιγότερο από ποτέ. Και δυστυχώ η ανθρωπιστική βοήθεια δεν μπορεί να λύσει όλα αυτά τα προβλήματα. Πιστεύω ακράδαντα τέλο, αλλά εξίσου σημαντικό, ότι Πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο να δημιουργήσουμε την σχέση, τη διασύνδεση μεταξύ ε, της ανάπτυξης και της ανθρωπιστικής βοήθειας υπό αυτά τις συνθήκες για να διοχετεύουμε τους πόρους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν θα εκπλαγείτε να ακούσετε ότι θα τελειώσω με ένα ευχαριστώ στις κυβερνήσεις σας για τη βοήθεια που μας παρέσχουν στην ανθρωπιστική, στον τομέα του προπολογισμού ανθρωπιστικής βοήθειας, διότι οι πληρωμές αυτές ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις στα πλαίσια του τακτικού προπολογισμού. Η ανθρωπιστική βοήθεια σώζει ζωές. Αν δεν έχουμε τα χρήματα, χάνουν τη ζωή τους οι άνθρωποι. Και είναι ένας τομέας όπου η δράση είναι άμεση. Δεσμευόμαστε σήμερα, πληρώνουμε αύριο. Συνεπώς, ελπίζω θα καταλάβετε ότι θα υπάρξουν οι πληρωμές ε, για να καλυφθούν οι ανάγκες και ε, ο προϋπολογισμός το 2015 θα καλύψει το κενό ανάμεσα στις δεσμεύσεις και τις πληρωμές. Διότι δεν πρέπει να λείψουν τα χρήματα σε αυτόν τον τομέα. Επ' αυτού θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δώσατε. Μ' αρέσει η δουλειά μου, αγαπώ τη δουλειά μου νομίζω ότι κάνω την καλύτερη δουλειά στην Επιτροπή και αγαπώ πολύ το προσωπικό μου. Μερικά από τα στελέχη μου βρίσκονται εδώ. Είναι καταπληκτικοί πρεσβευτές της Ευρώπης. Παρακαλώ να τους βοηθήσετε. Ε, Κύριε Επίτροπε, είναι η πρώτη φορά που προεδρεύω σε αυτή την Επιτροπή και μέχρι τώρα δεν ε, είχα ασχοληθεί με την ανθρωπιστική βοήθεια. Πιστεύω όμως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μία εξαιρετική πρέσβυρα. Ε, φαίνεται ξεκάθαρα ότι αγαπάτε τη δουλειά σας και ότι έχετε πάθος για αυτό που κάνετε. Και είναι εκπληκτική η δουλειά που κάνετε. Δηλαδή, κοιτάξτε εκεί το, την κλίμακα της ε, κρίσης. Τα έχετε δει αυτά με τα ίδια τα μάτια σας. Τι σημαίνει δηλαδή να ζει κάποιο σε μια χώρα που πλήττεται από την κρίση και πόσο προσπαθείτε να κάνετε ό,τι μπορείτε. Όπως είπατε κι εσείς, δεν μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα, έχουμε όμως κάποιες ευθύνες και πρέπει λοιπόν αυτές να τις αναλάβουμε στον υπερπολογισμό του 2014. Και πράγματι, ψηφίσαμε για να εξισωθούν, να εξισορροπήσουν οι πληρωμές ε, με τις ε, υποχρεώσεις. Όμως αυτό φυσικά είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής Προπολογισμών, Μα αφορά όμως και εμάς πάρα πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο στους ευρωβουλευτές και θα ήθελα πρώτα να μου πείτε ποιο από εσάς επιθυμεί το λόγο. Μας έχουν μείνει 15 λεπτά ακόμα και δεν ξέρω ποιοι θέλετε να μιλήσετε και πώ θα ε, χωρίσουμε το χρόνο. Ε, βλέπω ο κύριο Νόιζερ θέλει το λόγο, ο κύριο Στίερ, η κυρία Χαούτελα και η κυρία Χόιτεμποκ. Άλλο κανεί, άλλο ένα. Έχουμε περίπου τρία λεπτά για τον κάθε ένα από εσά και μετά θα δώσουμε το λόγο στην Επίτροπο για να απαντήσει. Α, και η κυρία Τόιερ. Μάλιστα. Μετά από τις ερωτήσεις σας θα ακούσουμε την Επίτροπο. Κύριε Νόιζερ, αρχίζετε, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε Γεωργίευα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την δουλειά που έχετε κάνει κατά τη διάρκεια της θητείας σας. Για μας ήταν μεγάλη ευχαρίστηση ε, που συνεργαστήκαμε. Και στην Αμερική υπάρχει μία έκφραση για εκείνους που δεν ασχολούνται και πολύ με τη δουλειά τους. Ε, τους λένε ε, κουτσές πάπιες, lame εντάξει, αλλά εσείς δεν είστε τελείως διαφορετικό από αυτό. Θα θέλαμε λοιπόν να σας ευχαριστήσουμε για τη δουλειά που έχετε κάνει και την αφοσίωση που έχετε δείξει κατά τη διάρκεια της θητείας σας και δεδομένων των πόρων που έχετε είναι και περιορισμένη η δύναμη του έργου σας. Πάρα πολλές κρίσεις έχουν οξυνθεί τα τελευταία χρόνια και δεν έχει παρατηρηθεί καμία αντίδραση στα κρατημέλη έτσι ώστε να αυξηθεί η χρηματοδότηση για την ανταπόκριση και την αντιμετώπιση τους. Και αυτό συνδέεται με τις διπλωματικές προτεραιότητες που υπάρχουν και με ορισμένα συγκεκαλυμμένα συμφέροντα. Ακούσαμε ορισμένους εκπρόσωπους των Ηνωμένων Εθνών και της Γενικής Διεύθυνσης ΕΚΟ και διαβάσαμε και τις εκθέσεις των γιατρών χωρίς σύνορα νωρίτερα. Και από όλα αυτά είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε υποτιμήσει τις συνέπειες της κρίσης στο Ιράκ, την Κεντρική Αφρική, το, Νότιο Σουδάν και ε, τις επιπτώσεις της πανδημίας του έμπολα και οι επόμενοι μήνες θα είναι πάρα πολύ δύσκολοι για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις κρίσεις. Τώρα, όσον αφορά τον έμπολα, η δική μας, η Επιτροπή θα ήθελε να ασχοληθεί περισσότερο με το πρόβλημα αυτό και να αυξηθεί η χρηματοδότηση για την καταπολέμηση του έμπολα και θα ήθελα λοιπόν να προωθήσω το θέμα αυτό για την ε, επόμενη ολομέλεια. Θέλουμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή της ε, καταπολέμησης του έμπολα, διότι αυτή είναι μια διακρατική απειλή. Είναι ευθύνη μας να αντιδράσουμε σε αυτή την απειλή που μπορεί να μην βρίσκεται ε, στο έδαφος μας, είναι όμως το κατόφλι μας. και οι συνέπειε είναι τώρα δραματικέ, θα είναι ακόμα περισσότερο δραματικέ όμω εάν επεκταθεί αυτή η κρίση. Πρέπει επίση να ε, προσπαθήσουμε να προασπίσουμε την ουδετερότητα και την αμεροληψία και η ανθρωπιστική βοήθεια να μην συνδέεται με τους πολιτικούς στόχους της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, τώρα θα ήθελα να ρωτήσω επίσης κάτι άλλο. Οι Φιλιππίνες ε, αυτή τη στιγμή πλήττονται από ε, χωρίς προηγούμενο φυσικές καταστροφές με τρομακτικές συνέπειες. Κάτι το οποίο δεν ε, ακούμε όμως πολύ συχνά στα μέσα ενημέρωσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να παρέχουμε ανθρωπιστική βοήθεια. Και θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω πώς ε, ανταποκρίνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε όλα αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Όπως είπε και ο σοσιαλιστής συνάδελφος, πιστεύω κι εγώ ότι αν θα έπρεπε να περιγράψουμε το έργο της κυρίας Επιτρόπου θα το περιγράφουμε ως ε, ηγετικό. Πραγματικά έχετε δείξει ηγετικό χαρακτήρα και έχετε συνεισφέρει πάρα πολύ στο, ότι, ε, στο να θεωρείται η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοπόρος στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Θα ήθελα λοιπόν και εγώ να συγχαρώ το έργο σας. πιστεύω πως ε, ένας από τους ε, λόγους ε, που έχετε αυτόν τον ηγετικό ρόλο ήταν, είναι ότι πραγματικά ήσασταν παρούσα οπουδήποτε υπήρχε ανάγκη. Εγώ θυμάμαι τι έγινε στην Κροατία, στη δική μου χώρα. Όταν πλημμύρισε η χώρα ήσασταν εκεί και δείξατε λοιπόν ηγετικό πρόσωπο. Γι' αυτό λοιπόν δεν εκπλήσωμε με το ότι σας στηρίζουν και οι περισσότεροι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρατε τώρα τη σημασία που έχει να φροντίσουμε ε, και να δώσουμε την δέουσα προσοχή σε προβλήματα και χώρες όπου ε, χρειάζεται. Για παράδειγμα στο Νότιο Σουδάν, το οποίο δεν φαίνεται και τόσο ε, πολύ τώρα τελευταία. Εγώ θα ήθελα να κάνω και μία πιο γενική ερώτηση. Όσον αφορά το ξέσπασμα του έμπολα, δόθηκε μεγάλη προσοχή τις τελευταίες εβδομάδες, η οποία βλέπω να υποχωρεί. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε εσείς πώς εκτιμάτε τις μελλοντικές εξελίξεις. Προς τα πού πηγαίνει δηλαδή η κατάσταση, ποιοι είναι οι πιθανοί κίνδυνοι και πώς μπορούμε να θέσουμε τον έμπολα υπό έλεγχο. Και μία άλλη ερώτηση πιο γενική. Δεδομένης της εμπειρίας σας, θα μπορούσατε να μας ε, πείτε πού βλέπετε να οδεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα χρόνια, ιδιαίτερα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής στην Τουρκία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Χάουτελα. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να σας συγχαρώ, κυρία Πίτροπε. Σας ε, πρωτογνώρισα κατά τη διάρκεια της ε, θητείας μου στο Συμβούλιο Ανάπτυξης και πραγματικά εκτιμώ πάρα πολύ τις ε, επιστολές που μας στέλνατε για τα ταξίδια σας στις περιοχές που αντιμετώπιζαν κρίση και την ε, ανταπόκρισή σας στις ανάγκες των περιοχών αυτών. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω και κατά την ε, παρουσίασή σας μας αναφέρατε σαφέστατα το πού βρισκόμαστε, το τι γίνεται στον κόσμο και το ότι πρέπει να δούμε και τις αιτίε που κρύβονται πίσω από τις ε, πρόσφατες ε, κρίσεις και να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις αιτίε. Η ερώτησή μου είναι παρόμοια με εκείνη του κυρίου Στίερ. Εσείς τι θα θέλατε να κληροδοτήσετε στην ε, επόμενη γενιά, στον επόμενο επίτροπο που θα αναλάβει το δικό σας χαρτοφυλάκιο όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια και εν ώψη της ε, συνόδου ε, στην Τουρκία. Στην Τουρκία. Και επίσης, ποια είναι τα έμπρακτα βήματα που έχουν γίνει για να συνδεθεί η ανθρωπιστική βοήθεια με την ε, στρατηγική, με την πολιτική και αν υπάρχει προθυμία ανάμεσα στους αρμόδιους φορείς να γίνει αυτή η σύνδεση, να ενώσουν αυτές τις γέφυρες. Σας ευχαριστώ. Θα θέλαμε τώρα να δώσουμε το λόγο στην κυρία Πίτροπο να απαντήσει και μετά να ακούσουμε τις επόμενες ερωτήσεις. Κυρία Πίτροπε, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Η αποφασιστικότητα που έχουμε δείξει προέρχεται από την ανάγκη που υπάρχει και πολλές φορές αισθάνομαι ότι η ανθρωπιστική βοήθεια είναι σαν το καναρίνι που είχαν οι ανθρακορίχοι στις ε, σύραγγες. Και εμείς είμαστε αυτό και είναι δική μας λοιπόν ευθύνη να ακρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου και να επιστήσουμε την προσοχή στο ότι υπάρχει ανάγκη και υπάρχουν ε, αιτίε που κρύβονται πίσω από τις κρίσεις. Και εδώ βρίσκεται και η ανησυχία μου ως προς αυτή την ψυχρή ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας της ε, κρίσης στην Ουκρανία η κρίση αυτή έχει προκύψει σε μια πάρα πολύ κακή χρονική στιγμή, σε μια στιγμή που χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ συλλογική προσπάθεια για να καταπολεμήσουμε τον εξτρεμισμό, για να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή. Θεωρώ πως τα κράτη-μέλη αντιδρούν πάρα πολύ καλά και κινητοποιούνται άμεσα όταν είναι σαφής η κατάσταση, όταν είναι σαφές το πρόβλημα. Αυτό το έχω δει πολλές φορές. Είναι όμως εξίσου σημαντικό να υπάρξει συντονισμός αυτής της κινητοποίησης. Και αυτό με μεταφέρει αμέσως σε μία από τις, ε, ένα από τα στοιχεία που πιστεύω πως ε, θέλω να κληροδοτήσω στον επόμενο επίτροπο. Αυτός ο μηχανισμός ανταπόκρισης σε έκτακτη ανάγκη. Είναι ένας ε, μηχανισμός που θα μας ε, ε, βοηθήσει να εντοπίσουμε και να ανταποκριθούμε άμεσα σε περιπτώσεις κρίσης και έκτακτης ανάγκης. Και όχι μία, πολλαπλές περιπτώσεις. Όταν το δοκιμάσαμε, είχαμε να αντιμετωπίσουμε πέντε κρίσεις ταυτόχρονα. Αυτός ο αριθμός θα πρέπει να αυξηθεί. Και θα πρέπει λοιπόν να είναι σημαντικό τόσο για τα κράτη-μέλη όσο και για εμάς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρειάζεται μια αξιολόγηση λοιπόν των, της κάθε περίπτωσης και μια συντονισμένη ανταπόκριση σε αυτές τις ανάγκες. Και έχει δίκιο ο κύριος ε, Νόιζερ όταν λέει ότι πολλές φορές αυτή η αντίδραση δεν είναι αρκετά γρήγορη. Θεωρώ ότι αυτό συμβαίνει ακριβώς εξαιτία του ότι υπάρχουν πολλές κρίσεις ταυτόχρονα στον κόσμο. Και δεν είμαστε καλά εξοπλισμένοι ως ε, κοινότητα για να ανταποκριθούμε σε πολλές κρίσεις ταυτόχρονα. Και όταν γίνεται κάτι τέτοιο, χάνουμε την μπάλα. Και καθοδηγούμαστε από τα μέσα ενημέρωσης και στρέφουμε την προσοχή μας όπου μας δείχνουν αυτά. Να πω όμως ότι εγώ και οι συνάδελφοί μου έχουμε δεσμευτεί για να διαθέσουμε το 50% των κονδυλίων μας για αυτό που λέμε ξεχασμένες κρίσεις, παραμελημένες κρίσεις. Και πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με το πώς θα κατανεμηθεί ο φόρτος εργασίας, πώς θα κατανεμηθεί αυτή η αντίδραση και ανταπόκριση και συντονισμός στην κρίση, έτσι ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Τώρα, όσον αφορά τις ερωτήσεις σε πολλών από εσάς για τον έμπολα. Να σας πω πως δυστυχώς δεν είμαι αισιόδοξη και πιστεύω πως δεν έχουμε δει ακόμα τις χειρότερες πτυχές αυτής της κρίσης. Και τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις ε, εκλεπτισμένες δυνατότητες που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε πιο επιθετικά την κρίση και να εντοπίσουμε τα κέντρα της. Υπάρχει ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας και μπορούμε να ζητήσουμε να αναπτύξει εξειδικευμένες δυνατότητες. Όμως υπάρχει μία διστακτικότητα και αυτό το καταλαβαίνω εν μέρη, διότι πολλοί θα πούν τι δουλειά έχει ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας με τον έμπολα γιατί ο έμπολα δεν έχει έρθει ακόμα σε εμά. Όμως, επαναλαμβάνω, πρέπει να είμαστε πιο επιθετικοί στην αντίδρασή μας, να είμαστε εκεί. Χρειάζεται να γίνουν περισσότερες επενδύσεις στην κατάρτιση περισσότερων ανθρωπιστικών οργανώσεων για την αντιμετώπιση του έμπολα, δεδομένης της κλίμακας που λαμβάνει και της έκτασης που λαμβάνει το ξέσπασμα αυτό. Προσπαθούμε και εμείς ε, λοιπόν να συνεργαστούμε με τους γιατρούς χωρίς σύνορα για την κατάρτιση περισσότερου προσωπικού. Όμως δεν φτάνουν τα μέσα που διαθέτουμε. Χρειάζεται να γίνουν περισσότερα με τα χρήματα που διαθέτουμε. Και πιστεύω πως όντως ήμασταν κάπως αργοί στην ε, αντίδρασή μας. Και χρειάζεται σε αυτές τις χώρες να γίνουν ε, μεγαλύτερες επενδύσεις στα συστήματα υγείας. Τοπικά, όχι μέσω ξένων επενδύσεων. Τώρα, όσον αφορά το τι μπορούμε να κάνουμε για να υπερασπιστούμε τις ε, αρχές μας αυτές, είναι να τις ε, τηρήσουμε. Να είμαστε συνεπείς. Όσον αφορά την ε, Ουκρανία, όταν η Ρωσία είχε στείλει την ανθρωπιστική βοήθεια πέρα από τα σύνορα, ήταν κάτι που ήταν αντίθετο προς τις αρχές που είχαμε. Όπως για παράδειγμα και στο Ιρακ πρέπει να φροντίσουμε αυτά που κάνουμε να είναι σύμφωνα με τις αρχές που θέλουμε να έχουμε και να συμφωνούν με αυτές. Και γιατί είναι σημαντικό να διατηρήσουμε λοιπόν αυτές τις αρχές, διότι μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτές ε, τις επόλεμες ζώνες μόνο όταν είμαστε ουδέτεροι. Και αυτό γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο. Ακριβώς όμως επειδή τα πράγματα γίνονται ολοένα και πιο δύσκολα, πρέπει να τηρήσουμε αυτές τις αρχές πιο αυστηρά. Όσον αφορά τις Φιλιππίνες, να σας πω ότι συνεχίζουμε τα προγράμματα που τρέχουν έχουμε πραγματικά παρατηρήσει αποκαρδιωτικές εξελίξεις. Μετά από τρία χρόνια η κρίση έχει ξεχαστεί. Και πάλι επιστρέφω σε αυτή τη δέσμευση που έχουμε αναλάβει για αυτό το ποσό των κονδυλίων που διαθέτουμε, το οποίο θα διατίθεται σε αυτές τις παραμελημένες κρίσεις. Παρατηρείται βέβαια κάποια ανάκαμψη και αυτό είναι ενθαρρυντικό ως προς αυτού του τύπου της κρίσης, όμως ε, χρειάζονται να γίνουν πολύ περισσότερα ακόμα. Ακριβώς όπως και στην ε, κρίση στην IT. Τώρα θα ήθελα να πω στον κύριο Στίερ ότι πραγματικά εκτιμούμε την, ε, το έργο της ε, ΕΚΟ, το έργο της ε, μας. Πραγματικά προσπαθούμε να είμαστε εκεί όπου υπάρχει ανάγκη και δεν μπορώ να τονίσω αρκετά την αξία που έχει η αλληλεγγύη, την αξία που έχει το να είμαστε δίπλα σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Τώρα, ως προς το πόσο φαίνεται το έργο μας, πιστεύω πως πρέπει να μας ρωτάτε πολύ πιο συχνά το τι κάνουμε για τις παραμελημένες περιπτώσεις. Να μας το υπενθυμίζετε. Και τώρα, όσο για το πού βλέπω να πηγαίνει η ανθρωπιστική βοήθεια, ποιο είναι το μέλλον, θα ήθελα να πω δύο πράγματα που συνδέονται και με τη δική μου κληρονομιά. Καταρχάς πιστεύω πως πρέπει να δεχτούμε το γεγονός ότι η ανθεκτικότητα είναι πάρα πολύ ε, σημαντική. Πρέπει να είμαστε ανθεκτικοί έτσι ώστε να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε και να μειώσουμε τις ε, ανθρωπιστικές κρίσεις στο μέλλον. Έπειτα, απολύτως απαραίτητο είναι να δημιουργηθεί σύμπνοια με τους ε, δωρητές, με τους χορηγούς από με τους, και νέους χορηγούς. Μπορεί να διαφωνούμε σε πολλά σημεία, όμως πρέπει να φροντίσουμε έτσι ώστε να δημιουργήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα κοινά σημεία. Και γι' αυτό έχω εντείνει τις επαφές με τις χώρες του κόλπου. Έχουν πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουν και τι είναι σημαντικό για εμάς. εμείς έχουμε την ε, τάση να ενεργούμε από θέση ισχύ, από κάποια θέση ανωτερότητας. Και γι' αυτό λοιπόν το λόγο πολλοί δεν μας, δεν μας υπολογίζουν, διότι θεωρούν ότι τους ε, αντιμετωπίζουμε αφιψηλού. Έτσι έγινε και στην ε, περίπτωση με το Ιράκ. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δείξουμε σεβασμό Διότι, για παράδειγμα, στην περίπτωση του Ιράκ έχουν γίνει συνδιαλλαγές με τη Σαουδική Αραβία και το ότι πρέπει να είμαστε διαλλακτικοί δεν σημαίνει ότι υποτασσόμαστε σε κάποιον άλλο. Σημαίνει ότι δείχνουμε υπευθυνότητα, η οποία υπευθυνότητα είναι και προς το δικό μας συμφέρον και προς το συμφέρον εκείνων που ε, χρειάζονται τη βοήθεια. Και τέλος, η συμβουλή που θα έδινα στην ομάδα της ε, ΕΚΟ είναι ότι Πρέπει να είστε περήφανοι. Πρέπει να είστε περήφανοι και να ε, ξέρετε ότι η Ευρώπη είναι μία οντότητα που φροντίζει για το καλό. Και αυτό πρέπει να πάρετε και να το συνεχίσετε. Ευχαριστώ κύριε Πίτροπε. Ε, ε, φαντάζομαι ότι σας εκτιμά και το προσωπικό σας και κάνετε πολύ καλή δουλειά και εσείς και το προσωπικό σας. Έχω τέσσερις ακόμα ομιλητές. Η κυρία Χάουμπουξ καταρχάς και μετά ο κύριος Ζέλερ. Θα ήθελα να επιστρέψω στην κρίση για τον έμπολα. Είπατε μόλις τώρα ότι πρέπει να δημιουργήσουμε περισσότερες ε, δυνατότητες. Πρέπει να δημιουργήσουμε δηλαδή περισσότερες δυνατότητες ανταπόκρισης. Ποιες είναι αυτές οι δυνατότητες ανταπόκρισης. Ε, διότι χθε είχα μια συνομιλία με τον κύριο Ροντιέ από τους γιατρούς χωρίς σύνορα, τον υπεύθυνο της ε, των Ευρωπαίων για τον χωρίς σύνορα και οι δικές του εκτιμήσεις και απαιτήσει ήταν ότι χρειάζεται περισσότερο προσωπικό, χρειάζεται καλύτερη, ε, καλύτερη υποδομή. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσω και την δική σας άποψη. Αυτές οι υποδομές υπάρχουν στις ανεπτυγμένες χώρες, στις δυτικές χώρες. Υπάρχει, παράδειγμα, κατάλληλη υποδομή στον ε, στρατό. Ε, θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, έχουν έρθει γιατροί χωρίς σύνορα σε εσάς για να σας μιλήσουν για τις ανάγκες που έχουν και αν ε, ναι, ποια είναι η δική σας τάση και τι άποψη έχετε για το ότι πρέπει να δημιουργηθούν ενέργειες γέφυρες που θα ενώσουν ε, εμάς με αυτές τις χώρες. Πάρα πολλές εταιρείες δεν πετάνε στις χώρες που υπάρχουν κρούσματα. Όμως πρέπει να υπάρχει δυνατότητα σε όποιον έχει ανάγκη να εγκαταλείψει αυτές τις ε, περιοχές. Επίσης θα ήθελα να προσθέσω ότι με χαροποίησε πάρα πολύ αυτό που είπατε, ότι δηλαδή αυτή η κρίση θέλει και πολιτικές ε, λύσεις και πιστεύω πως αυτή είναι μεγάλη πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι καινούρια Ευρωβουλευτής και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ για το ότι το είπατε αυτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριος Τσέλερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και την κυρία Επίτροπο για την περιεκτικότατη παρουσίασή της και απάντησή της. Ε, βλέπω ότι έχετε άμεση απόλυτη επίγνωση των προβλημάτων οι κρίσεις και οι ένοπλες σειράξεις ε, πλέον στον κόσμο δεν γνωρίζουν σύνορα, αλλά βλέπουμε τώρα ότι επεκτείνονται σε ολόκληρες υπήρους. Βλέπουμε σε όλη τη Δυτική Αφρική, την Κεντρική Αφρική, Ανατολική Αφρική, στην Εγγύη και Μέση Ανατολή. Βλέπουμε λοιπόν αυτές τις ε, ζώνες, βλέπουμε ακόμα και τι γίνεται με αυτές τις ε, παγωμένε ε, παγωμένες σειράξεις στο Αζερβαϊτζάν, στην Αρμενία, προβλήματα τα οποία δεν έχουν ακόμα λυθεί. Σήμερα το πρωί ακούσαμε την παρουσίαση του Απεσταλμένου των Ηνωμένων Εθνών. Και έτσι όπως το κατάλαβα εγώ, μας είπε λίγο πολύ με διπλωματικό τρόπο ότι τα προβλήματα τα ξέρουν εκείνοι που μπορούν να τα λύσουν αλλά υπάρχουν τόσα πολλά συμφέροντα, τόσα πολλά αντικρουόμενα συμφέροντα που δεν μπορεί να ε, δημιουργηθεί η κατάλληλη θέληση για να επιληθούν αυτά. Πρέπει λοιπόν να δούμε όλα αυτά τα, όλες αυτές τις πτυχές μαζί για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε την σωστή στρατηγική. Και μιλήσατε για την ανθρωπιστική βοήθεια και πιστεύω ότι πραγματικά, όπως είπατε κι εσείς, η ανθρωπιστική βοήθεια είναι ένα τσιρότο το πάνω στην πληγή. Δεν ε, λύνει το πρόβλημα. Όμως, πολλές φορές ε, το, το τσιρό το αυτό, αντί να βοηθήσει την πληγή να επουλωθεί, την κάνει χειρότερα. Και αυτό το έχουμε δει και με αυτές τις μειονότητες στο Ιράκ οι οποίες εγκατέλειψαν τα χωριά τους και τώρα έχουν γίνει πρόσφυγες, έχουν καταφύγει σε στρατόπεδα προσφύγων και εξαρτώνται από ανθρωπιστική βοήθεια. Όμως τώρα πρέπει να γίνει η σπορά για το χειμώνα και δεν μπορούν να πάνε στα χωράφια τους. Και όταν έρθει ο χειμώνας αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μπορέσουν να ε, καλλιεργήσουν ε, ε, την Αιγή τους, δεν θα μπορέσουν εν τέλει να τραφούν και τότε θα είναι πολύ χειρότερη η καταστροφή που θα προκύψει τον επόμενο χρόνο από αυτήν που έχουμε παρατηρήσει τώρα. Και τι γίνεται στην περιοχή αυτή. Οι μεν δίνουν όπλα γιατί πιστεύουν ότι αυτές οι μικρές ομάδες θα επωφεληθούν, οι άλλοι οδηγούν τους πρόσφυγες σε στρατόπεδα προσφύγων. Αυτό όμως που πρέπει να δούμε είναι τι θα γίνει όταν ενωθούν αυτά τα προβλήματα στο μέλλον. Ποιο θα είναι το μέλλον της χώρας αυτής. Βλέπουμε τι γίνεται ε, τώρα στο Νότιο Σουδάν με το δημοψήφισμα. Το δημοψήφισμα που έγινε για την ανεξαρτησία οδήγησε σε μαζική εφορία και χαρά. Όμως δεν έλυσε τις ε, διαμάχες που ε, υπάρχουν. Διαμάχες που είναι εθνικές, που είναι πολιτικές. Και διαμάχες αυτές δεν πρόκειται να σταματήσουν και στο μέλλον. Και βλέπουμε ότι καμία αποστολή, είτε αυτή είναι των Ηνωμένων Εθνών, είτε αυτή είναι των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν μπορεί να δώσει κάποια ικανοποιητική λύση στο πρόβλημα. Δεν μπορεί να ρυθμίσει την ε, κρίση, διότι δεν υπάρχει ασφάλεια στην περιοχή αυτή. Και τι γίνεται τώρα στο Νότιο Σουδάν, αρχίζει σε λίγο η περίοδος των βροχών και θα είναι ε, το έδαφος αυτό απροσπέλαστο για οποιονδήποτε θέλει να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια. Υπάρχει, θα ήθελα επομένω να ρωτήσω, ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή η πειθαρχία έτσι ώστε να ενωθούν τα κράτη-μέλη, να συνεργαστούν και να δώσουν μαζί κάποια λύση, να δημιουργηθεί μια από κοινού ε, στρατηγική, έτσι ώστε να αποφύγουμε περαιτέρω κλιμάκωση της κατάστασης. Πιστεύω ότι αυτά που μας είπατε ε, καθιστούν σαφές ότι είσαστε ένα από τα πρόσωπα τα οποία πραγματικά ε, έχει κερδίσει χωρίς κανένα δισταγμό τη στήριξη αυτού του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ κυρία Τόγια και μετά ο επόμενος συνάδελφος. Ναι, έχω μία ερώτηση, ένα αίτημα και μία προσωπική ερώτηση στη συνέχεια. Η πρώτη ερώτηση μου είναι η εξή. Εσείς είπατε ότι πρέπει να υπάρχει μια σχέση μεταξύ ανθρωπιστική βοήθειας και ανάπτυξης. Αν μπορείτε να μας δώσετε κάποια υπόδειξη ε, στο τέλος αυτής της τόσο έντονης δραστηριότητάς σας στη διάρκεια της θυσίας σας για κάτι τόσο δύσκολο αλλά και απαραίτητο. Το αίτημά μου είναι ε, όταν αναλάβατε τα νέα σας καθήκοντα να μην ξεχάσετε όταν θα αρχίσετε να νιώθετε μόνοι και βρεθείτε ενώπιον κρίσης να πείτε ότι αν η Ευρώπη είχε κάνει το τάδε στο περιβάλλον για παράδειγμα μην ξεχάσετε λοιπόν την ανάγκη να άρουμε όλα αυτά τα προβλήματα ακόμα και με νέα καθήκοντα. Όταν διαπιστώνει κάποιο ότι είναι η κρίση πρώτων πριλών, πριν προλάβει να σκάσει ανθρωπιστική βόμβα, ε, μήπω πρέπει να κάνει κάτι. Και θα ήθελα να σα κάνω και μια προσωπική ερώτηση. Είχατε χρόνο να ε, μάθετε γαλλικά στα τελευταία αυτά πέντε χρόνια. Σα θυμάμαι εδώ στην πρώτη σα ακρόαση πριν από πέντε χρόνια. Ήταν πολύ συγκινητική και πολύ έντονη. Όλου μα εξέπληξε. Σα χειροκροτήσαμε στο τέλο και είπατε ότι θα μαθαίνατε γαλλικά ε, βρήκατε χρόνο. Αν δεν βρήκατε χρόνο βέβαια είστε καθόλου δικαιολογημένοι. Καλύτερα με ονομάζεις Παύλο. Το, το επώνυμό μου είναι πολύ δύσκολο. Είμαι ο Παύλο για όλους σας. Πιο απλό. Πρώτα απ' όλα, εξ ονόματος όλης ομάδος, θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μας για την εξαιρετική δουλειά της Επιτρόπου. Παρακολούθησα τις δραστηριότητες σας από κοντά. Έχω δύο ερωτήματα. Το ένα αφορά τον επιμερισμό της ευθύνης. Τι πιστεύετε, ποιες χώρες θα πρέπει να επομίζονται μεγαλύτερο μέλος του βάρους της ευθύνης σε σχέση ε, οι χώρες που δημιουργούν αυτές τις κρίσεις ή εκείνοι που υποστηρίζουν αυτές τις χώρες. Μπορείτε να κατονομάσετε ορισμένες χώρες που θα μπορούσαν ή θα έπρεπε να δώσουν περισσότερα χρήματα. Δεύτερον, η ανθρωπιστική παρέμβαση, επέμβαση, βοήθεια χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν σε ορισμένε περιπτώσει με την άδεια του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΟΙΑ και σε ορισμένε περιπτώσει χωρί Στην κρίση της Ουκρανίας ακούστηκαν φήμες, εκτιμήσεις ότι πιθανόν η Ρωσία βρισκόταν από πίσω όσον αφορά το, την ανθρωπιστική βοήθεια παρέμβαση στην Ουκρανία. Πώς βλέπετε αυτή την ιδέα και ποιες είναι οι προοπτικές για το μέλλον πιστεύετε σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται αυτές οι δικαιολογίες ε, όταν γίνονται τέτοιου είδους παρεμβάσεις, στρατιωτικές δηλαδή. Και εγώ έχω μια ερώτηση για τον προπολογισμό. Αναφερθήκατε στα δημοσιονομικά προβλήματα για την ανθρωπιστική βοήθεια. Από ό,τι καταλαβαίνω, ζητήθηκαν επιπλέον 250.000 ευρώ, αλλά το θέμα παραμένει εκρεμές. Δεν ξέρουμε αν θα δοθούν, αν θα περιληφθούν στο προπολογισμό του 2015 ή θα υπάρξει περικοπή αυτού του ποσού. Και πώς επηρεάζεται η ανθρωπιστική βοήθεια στην πράξη. Πολύ σοβαρά ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα, για την ικανότητα απόκρισης ε, στην ε, επιδημία της έμπολα. Εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι να υπάρχει εξοπλισμός και παραγιατρικό προσωπικό. Δηλαδή σκηνές, νοσοκόμες και εξοπλισμός, όποια σειρά και αν πάρετε. Τώρα προσεγγίζουμε το στρατητικό προσωπικό για να δούμε κατά πόσον το στρατικό προσωπικό μπορεί να βοηθήσει ώστε να υπάρχουν σκηνές, εξοπλισμός και πιθανόν παραγιατρικό προσωπικό, νοσοκόμες δηλαδή όπως είπαμε, ε, ποιες είναι οι ικανότητες πολιτικής προστασίας των κρατών μελών. Και από ό,τι έχω καταλάβει πάλι, πολλές χώρες είτε έχουν είτε έχουν πολύ περιορισμένα μέσα και τις περισσότερες φορές ε, δεν τα μοιράζονται με το στρατηγικό. Γι' αυτό πιστεύω ότι η προσπάθειά μας θα έχει θετικά αποτελέσματα. Τώρα, τα πολλαπλά σημεία της κρίσης, κύριε Ζάιλερ. αν αρχίσουμε να βλέπουμε την κάθε κρίση ξεχωριστά, κάθε θερμό σημείο στον πλανήτη, θα φτάσουμε τα μεσάνυχτα. Διότι δυστυχώς υπάρχουν πολλές αιστείες αυτή τη στιγμή και βεβαίω που δεν συγκρίνονται με το μέγεθος που παρουσιάσαμε στο χάρτη, αλλά που θίγουν τους πληθυσμού. Εδώ αναφέρουμε τις σημαντικότερες κρίσεις. Προφανώς η πολιτική βούληση μπορεί να οδηγήσει σε λύσεις. Η ανθρωπιστική βοήθεια είναι αναγκαία, σίγουρα, επειδή η διάσωση των ζώων είναι πολύ σημαντικές, διότι πέρα ε, από όλα σώζονται ζωές. Δημιουργείται χώρος για τον άνθρωπο ακόμα και όταν υπάρχουν οι χειρότερες συγκρούσεις. Και εμείς, Ευρωπαίοι, πρέπει να το κάνουμε όταν υπάρχουν εκατομμύρια που χάνουν τη ζωή τους. Γι' αυτό η ανθρωπιστική βοήθεια είναι ένα πολύτυπο μέσο ανάμεσα στα μέσα με τα οποία αντιμετωπίζουμε τις κρίσεις. Αλλά δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τη ρίζα του προβλήματος και δεν μπορούμε μόνοι να δώσουμε πολιτικές λύσεις. Αυτή δεν είναι δουλειά μας. Δουλειά μας είναι, καθήκον μας είναι να δημιουργήσουμε χώρο για τον άνθρωπο ώστε να υπάρχει ανθρωπιά, να είμαστε άνθρωποι. Αυτός είναι ο στόχος τον οποίο πρέπει να επιτύχουμε. Δηλαδή, να τονώσουμε το στοιχείο του ανθρώπου και πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να δημιουργήσουμε ένα χώρο ανθρωπιάς. Για το Ιράκ ανησυχώ ειλικρινά. Τι θα γίνει αυτό το χειμώνα. Όταν ήμουν εκεί η θερμοκρασία είχε φτάσει στους 56 βαθμούς, αλλά σύντομα θα πέσει στους 0 βαθμούς και κάτω από το 0. Αλλά σας διαβεβαιώνω ότι ε, στην ανθρωπιστική κοινότητα δεν μας απασχολεί μόνο το να βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Σκεφτόμαστε όμως πώς η δράση μας μπορεί να περιορίσει το μέγεθος της κρίσης. Για παράδειγμα, όταν βρισκόμουν εκεί, με, λέγαμε τις κουρδικές αρχές, η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα δώσει περισσότερα μέσα για να ε, καθαριστούν οι νάρκες. Γιατί, διότι ακόμα και ε, όταν απελευθερωθούν χωριά, από πίσω ε, υπάρχουν οι νάρκες, υπάρχουν παγίδες. Αν θέλουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο να πάει σπίτι του, υπάρχει αυτή η προτεραιότητα, πρέπει να καθαρίσουμε το χώρο. Να καθαρίσουμε το χώρο από τις νάρκες. Γι' αυτό προσπαθούμε να βοηθήσουμε ε, στην επιστροφή των ατόμων. Αλλά αυτός ο συνδυασμός ε, των μέτρων που λαμβάνουμε ε, στο, στον τομέα της ασφάλειας είναι εξίσου σημαντικό με τα μέτρα που λαμβάνουμε στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Δεν μιλάω για το στρατιωτικό σκέλος, δεν είναι το δικό μας ε, δικός μας τομέας. Όταν όμως αρχίζουν να επιστρέφουν τα άτομα στα σπίτια τους, θα πρέπει να περιορίσουμε τους κινδύνους και να ανακουφίζουμε τον πόνο τους. Γενικότερα λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι πρέπει να επισημαίνουμε τα λάθη και την κακή συμπεριφορά. Πρέπει να ξέρουμε τι γιορτάζουμε. Γιορτάζουμε τη δημιουργία ενός κράτους. Μερικές φορές είναι ψευής πόθη αυτή. Δηλαδή, δεν μπορούμε να κάνουμε χειρουργικές επεμβάσεις, να αφαιρούμε αυτά που δεν θέλουμε. Πρέπει να κάνουμε λογικές εκτιμήσεις και αναφέρομαι στο Νότιο Σουδάνα και όχι μόνον. Δεν σας κάλυψα πλήρως σχετικά με το πώς αναπτύσσουμε σχέσεις μεταξύ ανθρωπιστικής βοήθειας και ανάπτυξης. Αυτό το οποίο κάνουμε στην πράξη είναι το εξής. Πρώτον, σε ευαίσθητα περιβάλλοντα προγραμματίζουμε ανθρωπιστική βοήθεια και παρεμβάσεις για την ανάπτυξη από κοινού. Και υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στην κοινή μας δράση. Και δεύτερον, σήμερα, περισσότερο από πριν από μερικά χρόνια, εφαρμόζουμε αυτή την έννοια των συγκριτικών πλεονεκτημάτων. Η ανθρωπιστική κοινότητα έχει ένα ε, συγκριτικό πλεονέκτημα ότι είναι παρούσα σε αυτές τις επικίνδυνες ζώνες. Υπάρχει μεγαλύτερη ανοχή όσο στην ασφάλεια. Οι εμπειρογνώμονες στον τόπο της ανάπτυξης, ε, περιοχές όπως η αυτή του Ελφαντοστού και αλλού ε, βοηθούν και εξασφαλίζουν μια σύνδεση ανάμεσα ε, στα μέσα αποκατάστασης και στην ανάπτυξη. Και δεύτερον, λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα για να κάνουμε συλλογή κονδυλίων εράνους σε γενικότερη βάση. Αλλά ε, επίσης στραφήκαμε στην Παγκόσμια Τράπεζα και στις Τράπεζες Αφρικανικής Ανάπτυξης ε, ζητώντας τους βοήθεια για να υπάρχει κάλυψη όλων των αναγκών. Καταλαβαίνω πολύ καλά τα γαλλικά, πρέπει να σας πω. Με μεγάλη χαρά ε, ακούω τα γαλλικά, είναι θαυμάσια γλώσσα. Καταλαβαίνω πολύ καλά, δεν μιλώ καλά τα γαλλικά. Προτιμώ λοιπόν να εκφράζομαι στα αγγλικά, δυστυχώς, για τα μέλη του Κοινοβουλίου που είναι γαλλόφωνοι. Ο επιμερισμός των ευθυνών του βάρους. Ποιος πρέπει να κάνει περισσότερα. Προφανώς πρέπει να ξεκινάμε από την αρχή ότι περισσότερη δουλειά σημαίνει περισσότερη ευθύνη. Λοιπόν, οι χώρες που αναπτύσσονται θα πρέπει να αναλάβουν, να δεσμευτούν να κάνουν περισσότερα. Είμαστε το 3% της παγκόσμιας οικονομίας στον κόσμο, αλλά 50% προς την ανθρωπιστική βοήθεια. Διότι καθώς ανεβαίνει η Κίνα και η Ρωσία, η Ρωσία κατεβαίνει. Εν πάση περιπτώσει δεν ήταν καλό παράδειγμα να το αναφέρω σήμερα. Αλλά καθώς αναπτύσσονται οι χώρες και γίνονται πιο πλούσιες, πρέπει να προσφέρουν και περισσότερα. Επίσης, οι κυβερνήσεις των χωρών πρέπει να κάνουν περισσότερα. Τουλάχιστον να προβλέπουν την πρόσβαση, αν δεν έχουν τα χρήματα, ας αφήσουν τη βοήθεια να φτάνει στους ανθρώπους που την έχουν ανάγκη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μία χώρα επιβεβαιώνει την κυριαρχία της. Όταν όμως υποφέρουν οι άνθρωποι, ε, αυτό δεν είναι απόλυτο αυτό, πρέπει να αλλάξει. Τώρα, η ανθρωπιστική βοήθεια πώς θα περάσει. Νομίζω ότι πρέπει το Συμβούλιο Ασφαλείας να δώσει τη σφραγίδα του, την έγκρισή του. Όπως ξέρετε υπάρχουν έξι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται και μεταξύ αυτών είναι να υπάρχει ένα περιβάλλον όπου αισθανόμαστε εμείς ότι υπάρχει αποδοχή αποδοχή της ε, βοήθειας, είτε πρόκειται για ανθρωπιστική είτε όχι. Αυτού του ίδιου η επέμβαση, πρέπει να πισθούν οι άνθρωποι ότι αυτού του ίδιου η επέμβαση βοηθάει και δεν είναι επιβλαβής. Νομίζω ότι εμείς κάνουμε προσεκτική ανάλυση όταν περνάμε τα σύνορα, διότι αν θέλετε το να περάσουμε τα σύνορα χωρίς να έχουμε την έγκριση είναι η τελευταία εσχάτη προσφυγή μας. Και σας διαβεβαιώνε ότι μετράω τα δάχτυλά μου λιγότερες από πέντε φορές είναι εκείνες που το κάναμε αυτό. Γιατί? Διότι από τη στιγμή που διατρέχετε τέτοιους κινδύνους ανοίγεται ε, την πόρτα και σε άλλους να το κάνουν. Ε, τώρα για ε, τη Ρωσία για παράδειγμα λένε πολύ καλά εσείς θα πάτε, πήγατε στη Συρία, θα πάμε στην Ουκρανία. Βλέπετε τι γίνεται. Αλλά σημειωτένω ότι για τη Συρία υπήρχε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας που είχε πει ότι πρέπει να σωθούν οι ζωές και συνεπώς μπορεί να πάει η ανθρωπιστική βοήθεια να περάσει τα σύνορα. Γι' αυτό νομίζω είναι πολύ δύσκολο και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν επεμβαίνουμε χωρίς να σεβόμαστε την κυριαρχία της κάθε χώρας. Τώρα, για τον προπολογισμό. Ο προπολογισμό. hopeful. Ελπίζω ότι θα πριτανεύσει η λογική. Νομίζω ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να αντιληφθούν ότι δεν είναι μόνο το σωστό, αλλά είναι προς το συμφέρον μας να βοηθήσουμε ώστε να μπορέσουμε να περιορίσουμε τις περιοχές σύραξης. Και η εντύπωσή μου είναι ότι υπάρχει κάποια τάση ε, χρηματοδότησης ε, των πιστώσεων πληρωμών για την ανθρωπιστική βοήθεια. Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, αυτό είναι εξαίρεση, για την ανθρωπιστική βοήθεια υπάρχει συμφωνία ε, αύξησης ε, των πιστώσεων πληρωμών στο επίπεδο των δεσμεύσεων. Και ξέρετε ότι οι διάφοροι ε, επίτροποι, ο καθένας προσπιζόταν το δικό του χαρτοφυλάκιο, αλλά τελικώς αποφασίσαμε να επικεντρωθούμε στην ανθρωπιστική βοήθεια και ελπίζω το αυτό να κάνουν και το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν χρειάζεστε κάποιον να παρακαλέσει στο πλάι σας, φωνάξτε με, θα είμαι εκεί. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Πραγματικά μας δώσατε ε, πράγματα να σκεφτούμε. Μας είπατε ότι αυτή είναι η χειρότερη κρίση από την κρίση των προσφύγων που είχαμε το 1945 και πραγματικά παρακολουθούσα ένα πρόγραμμα για την κρίση αυτή ε, το καλοκαίρι και τα εκατομμύρια των ανθρώπων που εκτοπίστηκαν. Κάποιοι έχετε ζήσει στην ιστορία και τα μαθαίνετε στην ιστορία. Σήμερα τα πράγματα είναι χειρότερα. Και καταφέραμε να φτάσουμε στους πολίτες. Ακούμε ε, Σύριους που, Σύρους που ζουν ε, στις γειτονικές χώρες ε, και ακόμα και για τις χώρες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της Ευρώπης είναι αδιανόητο το να φεύγουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Σήμερα το πρωί ε, εκπρόσωπος των ΗΕ Εθνών μας είπε ότι όλες αυτές ε, οι σειράξεις είναι ανθρωπογενείς και όντως είναι ανθρωπογενές. Ε, ε, υπάρχουν και γυναίκες που υπόκεινται τις συνέπειες αυτής της κρίσης και είναι πονίδιστο το γεγονός ότι δεν μας μαθαίνει τίποτα ιστορία κάνουμε κύκλους και προκαλούμε ακόμα περισσότερο πόνο στους ανθρώπους. Και το ερώτημα λοιπόν για όλους μας εδώ είναι τι σκοπεύουμε να κάνουμε από αυτού, τι ευθύνη έχουμε εμείς και το τελευταίο θέμα που θίξαμε είναι ο προπολογισμό και εκεί έχουμε ευθύνη. Υπάρχει μια κατάσταση στην οποία υπάρχει έτοιμα ε, να υπάρχουν περισσότερα χρήματα. Ε, θα μιλήσουν όλοι για την Ουκρανία, για τη Συρία, για το Ιράκ, για την κρίση του εμπόλα, για την... Ε, ε, τα προβλήματα στην ε, ε, Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής, αλλά πραγματικά πρέπει να αποδείξουμε εάν ε, πραγματικά εννοούμε ότι θα δώσουμε ανθρωπιστική βοήθεια. Πρέπει να προκαταβληθούν τα χρήματα, γιατί δεν έχουν σχέση με τις άλλες γραμμές του προπολογισμού. Ακούω πολλά στη χώρα μου για την Ευρωπαϊκή Γραφειοκρατία και το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να κατασπαταλά τα χρήματα, αλλά ξέρω μιλώντα σε υπαλλήλου και σε μη κυβερνητικέ οργανώσει ε, ότι χάνεται πολλής χρόνο προσπαθώντα να διοχετεύσουμε τα χρήματα ώστε να καλύψουμε τι δεσμεύσει μα. Αυτό είναι σπατάλη ενέργεια. Θα μπορούσαμε να είναι πολύ πιο αποτελεσματικοί και να δοπανούμε αυτά τα χρήματα με περισσότερη σοφροσύνη αν είχαμε περισσότερη ευχαίρεια στον προπολογισμό. Μα είπατε ότι θα έρχεται να παρακαλέσετε μαζί μα. Θα κάνουμε εμεί ό,τι μπορούμε στην Επιτροπή Προπολογισμών και στο Συμβούλιο, διότι νομίζω ότι όλοι επιθυμούμε να υπάρχει κατάλληλη χρηματοδότηση για την ανθρωπιστική βοήθεια και οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη να λαμβάνουν αυτά που χρειάζονται. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν ξέρουμε σίγουρα αν είναι η τελευταία φορά που θα έρχεστε στην Επιτροπή μας, αλλά σίγουρα Εκτιμώ το γεγονός ότι ήρθατε εδώ σήμερα και μας κάνετε μια τόσο καλή παρουσίαση της κατάστασης και χαίρομαι που υπάρχει κάποιος στο πλευρό μας, στο πλευρό της Ευρώπης που δίνει μάχη για την ανθρωπιστική βοήθεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν που ήρθατε εδώ σήμερα και είμαστε στη διάθεσή σας για συνεργασία με οποιαδήποτε ιδιότητα στο μέλλον. And now, um, that is the end of our business. Αυτό είναι το τέλος των εργασιών μας για σήμερα. Δεν μου έχει ε, δοθεί κάποια ενημέρωση για κάτι άλλο. Η επόμενη συνεδρίαση έχουμε τη Δευτέρα στις 4.30 με τον Επίτροπο Πίμπαλξ για να συζητήσουμε για το στρατηγικό διάλογο είστε επανειδήν ε, και η συνεδρίαση των συντονιστών για τους συντονιστέ, θα ξεκινήσει σε πέντε λεπτά. Για όλους όσους δεν συμμετέχουν στη συνεδρίαση των συντονιστών, ε, παρακαλώ να αποχωρήσετε από την αίθουσα και θα συνεχίσουμε με τους συντονιστέ σε πέντε λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ καλή συνεδρίαση σήμερα και ελπίζω να ήταν χρήσιμη και για σας.